I recall this has always been a problem in the previous years. Thank you very much. Thank you, Mr. Kukan. And now the floor to Mr. Manolis Kefalogiannis, Chair of the Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τα θέματα στην Τουρκία σε σχέση με την βία εναντίον των ε, γυναικών και των κοριτσιών δεν είναι σε καλό σημείο. Αυτό αποδεικνύεται και από στοιχεία τα οποία ε, παρουσιάστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου 38% των γυναικών έχουν δεχτεί σωματική σεξουαλική βία από τον σύντροφό του, 15% των γυναικών αναγκάστηκαν σε γάμο πριν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο δείκτης ανισότητας των φίλων για τη συγκεκριμένη χώρα είναι στη θέση 69. Ε, διεθνείς δείχτες ε, ε, έμφυλου χάσματος που μετράει το χάσμα βάσει των εκπαιδευτικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων έχουν κατατάξει τη χώρα στην 130η θέση και έρευνα του ίδιου του Υπουργείου Κοινωνικών Πολιτικών της Τουρκίας δείχνει ότι το 86% των γυναικών έχουν αντιμετωπίσει σωματική ή ψυχολογική βία από την οικογένειά τους και τους συντρόφους τους. Ε, η λύση είναι αυτή που είπε και ο κύριος Κούκαν όπως χρειάζεται τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι η πολιτική βούληση, ελεκτικοί μηχανισμοί για πρόληψη και καταστολή αυτής της βίας, ενημέρωση των κοριτσιών σε αυτές τις χώρες και των γυναικών για τα δικαιώματά τους και η πρόσβαση σε νομική υποστήριξη και υπηρεσίες υγείας και στέρασης είναι πολύ μικρή η συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε αυτή τη χώρα, κυρίως για γυναίκες που εγκατέλειψαν τους συζύγους τους ή ε, βρίσκονται ανυπεράσπιστες για δικαιώματα τα οποία έχουν όλες οι πολιτισμένες χώρες του ειδικού κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ε,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 rekao naše stavove i naše pozicije. I treba reći da je i Albanija jedna od onih zemalja koja ima relativno dobar pravni sustav uz implementaciju Istanbulske konvencije i ostali, ostalo zakonodavstvo je relativno solidno. Međutim, naravno, kao što smo čuli od mojih kolega i kolegica, problem je u implementaciji. I problem je uopće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 problema nasilja, diskriminacije žena i tako dalje. 8% seksualnog nasilja. U gradskim četvrtima, u gradovima je ta situacija malo povoljnija. Ali naravno da nije dobra. I dobro je gospođa McGuinness rekla pa i mi u Europskoj uniji imamo takve probleme, pa mi u Hrvatskoj imamo takve probleme. Ne možemo, ne možemo si reći da nemamo, kad ih imamo. Ali je činjenica da zemlje na Zapadnom Balkanu ipak imaju većih problema. I u tom kontekstu mislim da je dobra ova rasprava i mislim da je vrlo važno da mi kao zastupnice i zastupnici permanentno ukazujemo na naše stavove i tražimo od vlada na zapadnom balkanu kad su to već zemlje kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje da implementiraju ono što su naši pravni propisi.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 Grazie. Signora Rotanen, two minutes.